Καλημέρα σε όλους. Buongiorno a tutti. Καλημέρα. Πρωτίστως θέλω να χαιρετήσω όλους τους παριστάμενους. Είναι πολύ ιδιαίτερη σημερινή ημέρα. Θέλω λοιπόν να χαιρετήσω όχι μόνο όλους ε, από την Επιτροπή Γεωργίας, αλλά και όλους τους παρόντες από τις διάφορες γεωργικές οργανώσεις όλης της Ευρώπης. Από την Κόπα Κοζέκα βέβαια, Πέκα ε, και βέβαια θέλω να χαιρετήσω τους προέδρους, τους Ιταλούς προέδρους των ε, γεωργικών συνεταιρισμών, τους Τζέπε Πολίτη και Φράνκο Περάσινα και όλους τους άλλους που είναι σήμερα παρόντες. Αγαπητέ Επίτροπε, σας ε, καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, όπως σε όλες τις άλλες περιστάσεις που έχετε έρθει εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας, να μας παρουσιάσετε την ε, εξαιρετικά ογκώδη πρόταση για την ε, νέα θητεία με την μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής. Η Επιτροπή, που η Επιτροπή ενέκρινε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Το Κοινοβούλιο είναι ο χώρος όπου υποσωπεύονται οι ευαισθησίες ε, των Ευρωπαίων πολιτών και μπορούν πραγματικά να εκφραστούν. Είμαστε πεπισμένοι ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει αυτή η πρώτη επίσημη ανακοίνωση και πληροφόρηση πάνω στις προτάσεις που ορίμασαν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις τις οποίες θα μας παρουσιάσετε, αγαπητέ Επίτροπε, συνέρχονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο και ιδιαίτερο σενάριο. Από τη μια πλευρά έχουμε όλη επίγνωση της πολύ ευαίσθητης στιγμής στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αγορές ε, όλο και πιο μεταβλητές, όλο και πιο ανταγωνιστικές και όλο και μεγαλύτερες έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ τον ε, ε, παραγωγικό ιστό της Ευρώπης από βορρά σε νότο και από δύση ανατολή γνωρίζουμε τι θα σήμαινε μια ε, απομείωση του δικού μας ε, παραγωγικού αντιμετωπίζονται Αντιμετωπίζονται τις δύο μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει ε, η Ευρώπη της ασφάλειας, της ψηφιστικής ασφάλειας αφενός και του περιβαλλοντικού ρόλου και κοινωνικού ρόλου εκατομμυρίων γεωργών που σήμερα κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ήπεθρο. Είναι δύο πολύ μεγάλες προκλήσεις που οι δύο εκθέσεις που υιοθετήθηκαν σε αυτή την Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Ζωνς Λάιον και Άγιον Τες έχουν τύχει πολύ μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια και έχουν απομονώσει ακριβώς αυτές τις δύο προκλήσεις ως ύψιστες προτεραιότητες. Μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση που θα μπορέσει πραγματικά να γεφυρώσει δύο κατά φαινόμενα συμφιλίωτες προκλήσεις, δηλαδή μεγαλύτερη παραγωγή αλλά με λιγότερη ρήπανση. Ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει αηφορία, περιβαλλοντική αηφορία, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να έχουμε εγγυηθεί την οικονομική αηφορία των γεωργικών επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε ότι από αυτή την πτυχή σήμερα η κίνδυνη είναι πολύ πιο συχνή και πολύ ευρύτερη και ενδονότερη από το παρελθόν. Είμαστε ενώπιον μιας μεταρρύθμισης εκπληκτικής ε, σημασίας και εμβέλειας που θα συνοδεύσει τους γεωργούς μας σε μια νέα εποχή όπου το ευμετάβλητο θα γίνει πλέον συστηματικό φαινόμενο και επομένω οι γεωργοί θα έχουν ανάγκη νέων εργαλείων για να μπορέσουν να χειριστούν μια αναπόφευκτη όσο και δύσκολη κατάσταση. Σα υπενθυμίζω ότι αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό ε, δοκιμαστικός, ε, ε, δοκιμαστικό εργαστήριο, αν θέλετε, και σε θεσμικό επίπεδο. Για πρώτη φορά η μεταρρύθμιση ε, της κοινή αγροτική πολιτικής επισέρχεται στη διαδικασία τη συναπόφευση. Και αυτό συνεπάγεται πολύ σημαντική ευθύνη. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε, όπως ήδη αποδέχθηκε σε προηγούμενες περιστάσεις, να εκπονήσουμε πολύ σημαντική εργασία, χρήσιμη και για τους γεωργούς μας, αλλά και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Επίτροπο που ήρθε άμεσα ανταποκρινόμενος εδώ στην, Ευρωπαϊ... στην Επιτροπή Γεωργίας και δίνοντάς του τον λόγο τον πληροφορώ πρωτού ξεκινήσει η σημαντική αυτή συζήτηση, ότι είναι πολύ περιορισμένο ο χρόνο μα, ότι ο επίτροπο θα πρέπει το αργότερο να αποχωρήσει το 12.30. Εν θα ακολουθήσω βέβαια τη διαδικασία που πάντα έχουμε ακολουθήσει, δίνοντα το λόγο αμέσω μετά την εισήγηση του Επιτρόπου στου συντονιστέ των πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια στον εισηγητών πάνω στη μεταρρύθμιση και σε οποιοδήποτε στη συνέχεια άλλο βουλευτή που ε, θα υποβάλει σχετικό αίτημα. Ο επίτροπο μου είπε επίση, ότι τις επόμενες ώρες θα αποσταλεί σε, μέσω email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής τα πλήρη και επίσημα, το πλήρες και επίσημο κείμενο της πρώτας μεταρρύθμισης. Εάν δεν υπάρχουν ε, ε παρεμβάσεις επί διαδικαστικό, δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Θα έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε. Διαφορετικό δεν τα καταφέρουμε. Τάσαν Τσόλος λοιπόν. Έχετε το λόγο. Euh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, είχα έρθει πριν από ένα περίπου χρόνο ε, ενώπιόν σας με τις ακροάσεις για την μεταρρύθμιση την οποία είχα χαρακτηρίσει ως κύριο και κατά προτεραιότητα στοιχείο της εντολής που αναλάμβανα. Έχουμε λοιπόν μετά την έγκριση της Επιτροπής από την Επιτροπή των Προτάσεων αυτών έρχομαι ενώπιον σας να σα παρουσιάσω αυτέ τι προτάσει, Οπότε τι είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, όχι σε επόμενε ώρε, αλλά στα επόμενα λεπτά θα ε, φτάσει στο ταχυδρομείο σα το ηλεκτρονικό, το σύνολο των προτάσεων που υιοθέτησε σήμερα η Επιτροπή στη συλλογική της μορφή και ασφαλώς επόμενες ε, ημέρες, εβδομάδες θα μπορέσουμε να συζητήσουμε λεπτομερέστερα τις προτάσεις αυτές είναι η πρώτη φορά που εσείς συμμετέχετε με την συναπόφαση πλήρως στην επεξεργασία του κειμένου αυτού. Φριστόμαστε λοιπόν σε, μια, σε ένα σημείο καμπής ως προς την πολιτική της Γεωργίας. Έγινε ο δημόσιος διάλογος, τον οποίο, του οποίου έθεσα ε, τα θεμέλια στις 12 Απριλίου 2010 εδώ. Η ανακοίνωση της Επιτροπής ακολούθησε τον Νοέμβριο του 2010. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την προστιθέμενη αξία που προσφέρατε εσείς σε όλο αυτό το διάλογο, μαζί με τη συμμετοχή σας στο δημόσιο διάλογο, με τις εκθέσεις Lion και Des, αλλά και γενικότερα με τη συμβόλη στις συζητήσεις μας. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο επαναπροσδιορισμός της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής ε, είναι απαραίτητος, και πρέπει να εξασφαλιστεί μια νέα ισορροπία μέσα σε μια πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ της κοινωνίας η οποία προσφέρει δημοσιονομικούς πόρους για να στηρίξει μια πολιτική όπως την κοινή γεωργική πολιτική και τους γεωργούς και των γεωργών που βρίσκονται στη βάση του οικοσυστήματος ε, και προσφέρουν, παράγουν το ε, σύνολο των διατροφικών μας αγαθών. Έτσι λοιπόν, στόχοι μας είναι να ε, καταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα υπηρέτη της ε, γεωργικής και διατροφικής μας ασφάλειας. Οικονομική λοιπόν και οικολογική προσέγγιση, προσέγγιση η οποία θα επιτρέψει την ε, ανάπτυξη κατά τρόπο εναρμονισμένο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γεωργίας και ένα στόχος οριζόντιος των οποίων πολλές ε, φορές έχουμε συζητήσει και θα πρέπει να δείτε κι εσείς, απλούστευση της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής. Πρώτος στόχος λοιπόν, ανταγωνιστικότητα όλων των ευρωπαϊκών γεωργιών, όλης της γεωργίας στην Ευρώπη για την διατροφική ασφάλεια. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προαχθεί με πολιτικές οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο και τις οικονομικές εξελίξεις μέσω δύο τομέων, δηλαδή των αγορών και του εισοδήματο των γεωργών. Οι ανησυχίες έχουν μετακυλιστεί από το απλό ζήτημα της ε, διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και έχουν περάσει πλέον στο ζήτημα, στο πρόβλημα της ε, αστάθεια των αγορών και της πτυτικότητα των τιμών και των εισοδημάτων. Για τη γεωργία λοιπόν της Ευρώπης το πρόβλημα δεν είναι μια φυσική καταστροφή, η αλλαγή του κλίμακος ή κάποια δυσμενή καιρικά φαινόμενα, αλλά η ραγδαία πτώση του εισοδήματος και των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Επανέρχεται πάντα το ζήτημα λοιπόν του εισοδήματος των γεωργών που έχει υποβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και κατά τρόπον που δεν έχει αντιμετωπίσει κανένας άλλο οικονομικός τομέας. Τι απάντηση μπορούμε να δώσουμε σε αυτό το ζήτημα, του εισοδήματο δηλαδή. Πρώτον, νέε άμεσε πληρωμέ. Η αποτελεσματικότητα τη πολιτική μα έχει υποβαθμιστεί. Οι άμεσες πληρωμές με το παλαιό του σύστημα και την ιστορική αναφορά έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους, αποδυναμώνονται δε από την έλλειψη αξιοπιστία και διαφάνεια σε σχέση με το ευρύτερο κοινό. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν επιλογέ οι παλές ιστορικές αναφορές έχουν ξεπεραστεί και πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα νέο, πολύ πιο εστιασμένο, που να έχει να κάνει με τις επιφάνειες και έτος αναφορά το 2014. Η γεωργική ε, επιφάνεια η οποία θα αξιοποιηθεί θα είναι ένα νέο στοιχείο. Θα λαμβάνεται υπόψη και η παραγωγική διάσταση και η έννοια του δημοσίου αγαθού που παράγεται από την εν η επιφάνεια. Η δε προσέγγιση αυτή σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς τη σύγκληση. Γιατί η ίδια παραγωγικότητα, το ίδιο επίπεδο παραγωγής δημόσιου αγαθού σημαίνει ταυτόχρονα και ισότιμο επίπεδο στήριξης. Γιατί λοιπόν περιορίζουμε τη σύγκληση στο 1 τρίτο της διαφοράς μεταξύ της χαμηλότερης πληρωμής και το 90% του μέσου όρου ανά την Ευρώπη κατά την ε, δημοσιονομική περίοδο. Όπως γνωρίζετε, κυρία γεωργική πολιτική προχωρήσαμε τα ταυτόχρονα παράλληλα με τι συστήσει για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Πράγμα το οποίο είχαμε πολύ καιρό να δούμε στη δικασία μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Πρέπει λοιπόν οι στόχοι μα βεβαίω να ληφθούν υπόψη, αλλά ταυτόχρονα ληφθεί υπόψη και η δημοσιονομική η δυνατότητα ε, αντοχή αυτών των στόχων. Πόσο εφικτή είναι η στόχη αυτή δηλαδή με τα δημοσιονομικά δεδομένα που διαμορφώνονται τώρα. Αυτό σημαίνει να μετρήσουμε τι είναι δυνατόν και να δώσουμε σωστές ισορροπίες. Και πάνω απ' όλα να δώσουμε όθηση προς την ορθή κατεύθυνση, πράγμα το οποίο καταφέρνουμε πιστεύω με τις άμεσες πληρωμές κυρίως και τις προσπάθειες για τη σύγκληση με τις νέες προτάσεις. Φτάνουμε λοιπόν σε μια πρώτη φάση μέχρι το 2020 και ορίζουμε στόχο πολύ πιο ισορροπημένο για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές. Για τα στοιχεία εσωτερικής σύγκληση στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες που δεν εξαρτώνται από εξωτερικούς δημοσιονομικούς παράγοντες αλλά που επίσης έχουν πολύ μεγάλη σημασία προσδιορίζουμε έναν ταχύτερο στόχο που θα κληθεί να είναι αποτελεσματικός για τις πληρωμές που θα καταβάλλονται από το 2019 δυνάμει του προϋπολογισμού του 2020. Στη συνέχεια διαφοροποιημένη στήριξη επί τη βάση των αντικειμενικών αναγκών που θα καταγράφονται. Η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της, ζωτικό, της βιωσιμότητας του γεωργικού τομέα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αντικειμενική διαφοροποίηση της στήριξης. Και γι' αυτό προτείνουμε στα κράτη-μέλη ένα μηχανισμό στήριξης άμεση, άμεσο, άμεση στήριξης και εξελικτικό μηχανισμό με βοήθεια προς τον νέο γεωργό όπου προτείνουμε να διατηρηθεί μέχρι το 2% των εθνικών κονδυλίων μια πρόσθετη πληρωμή που θα αντιστοιχούσε στο 25% του μέσου όρου των όσων δικαιούνται για ένα μέγιστο των 25 ε, εκταρίων ανά νέο γεωργό για τα πρώτα χρόνια. Πρόκειται λοιπόν για ένα διαρθρωτικό μέτρο το οποίο ανταποκρίνεται στις ε, δημογραφικές ε, προκλήσεις, πρόκληση δηλαδή για όλα τα κράτη-μέλη, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με την επιβίωση των ε, περιοχών της υπαίθρου και άρα αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι στην ε, διάθεση των κρατών μελών, μάλλον πρέπει να είναι υποχρεωτικός για όλα τα κράτη-μέλη. Μετά θα έχουμε τις συνδυασμένες ενισχύσεις, πρέπει να έχουμε το θάρρος να προχωρήσουμε έστω και ενάντια στο κύμα, ε, ενάντια στη μόδα των οικονομικών θεωριών ε, και να τις διακηρύξουμε ξεπερασμένως ήταν απαραίτητο για να ε, συντηρήσουμε, να προστατέψουμε τους ευάλωτους ε, τομείς. Έτσι λοιπόν προτείνουμε να διαφυλάξουμε αυτό το μηχανισμό υπό την προϋπόθεση όμως ότι κάθε χρήση των συνδυασμένων πληρωμών θα είναι αιτιολογημένη. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να εστιάσουμε στα κράτη-μέλη κατά 5% της ενισχύσεις που προτείνει ο πρώτος πυλώνας προς στήριξη της γεωργίας που βρίσκεται σε υποβαθμισμένες ή λιγότερο πλεονεκτικές ζώνες. Αυτό σημαίνει και, αυτό γίνεται μάλλον και για λόγους περισσότερης ε, δικαιοσύνης, ισότητας δηλαδή, αλλά και για να συμβάλλουμε στην ε, διατροφική ασφάλεια και έτσι εξασφαλίζουμε την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου στις περιοχές αυτές τις λιγότερο πλεονεκτικές με ένα μέγιστο της ενίσχυσης στα 300 ευρώ ανά εκτάριο. Και έτσι εξασφαλίζουμε την κινητικότητα του παραγωγικού κεφαλαίου οπουδήποτε και αν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη γεωργία μας αλλά και για την ενίσχυση που θα δίνεται στο εισόδημα του γεωργού και στις δομές στις οποίες πραγματικά χρειάζεται. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω παρεπιπτόντως ότι μάλλον δεν χρειάζεται ενίσχυση ε, με, ε, με γεωργική στήριξη, δηλαδή ένα γήπεδο γκολφ ή ένα αεροδρόμιο Φερρυπίν. Και γι' αυτό είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε πολύ αυστηρό προσδορισμό του ε, ενεργού, δραστήριου δηλαδή γεωργού, με επακριβή κριτήρια, έτσι ώστε να μην βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση οι πραγματικοί γεωργοί, έστω και αν είναι μερικής απασχόλησης. Και γι' αυτό ε, ορίζουμε ένα κριτήριο βάσει των οποίων η άνεση ενίσχυση που χορηγείται θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 5% τουλάχιστον των μη γεωργικών ε, ε, εσόδων του ετούντος την ενίσχυση. Επίσης, προτιστορίζουμε και ελάχιστη προϋπόθεση γεωργικής εργασίας, γιατί βέβαια δεν μπορούμε να ενισχύουμε μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής τον γεωργό του καναπέ. Sofa Farmer. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφερθώ στο κατά πόσον είναι δυνατό να μιλούμε για ενίσχυση στη βάση του, εισοδήματο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σταδιακή μείωση των ενισχύσεων επί τη βάση ενό εισοδήματο που ξεκινάει στα 150.000 ευρώ με ανώτατο επίπεδο τα 300.000 ευρώ, πράγμα το οποίο αντιστοιχεί σε ε, ανησυχίε που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στην έκθεση DES τον Ιούνιο, ως προς τον κίνδυνο να αμφισβητηθεί η νομιμότητα των άμεσων ε, πληρωμών. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μηχανισμό ο οποίος ε, λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση στη γεωργία και δεν θέτει σε υποδέστερη θέση τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες δημιουργούν πραγματικά νέες θέσεις εργασίας. Το μισθολογικό, η μισθολογική βάζα, μάζα λοιπόν θα υπολογίζεται στο όριο θέση σε λειτουργία της ε, σταδιακής αυτής μείωσης. Και έτσι προχωρούμε με την ε, λήψη υπόψη και της καλής διαχείρισης των φυσικών πόρων που υπάρχουν. Δηλαδή έχουμε μια πράσινη βοήθεια η οποία δεν θα υποβληθεί στη σταδιακή μείωση, θα εξαιρεθεί τη σταδιακή μειώση. Θέλουμε επίσης να δώσουμε νέες βάσεις για ανταγωνιστικότητα, οικονομική και οικολογική ανταγωνιστικότητα της ε, νέας κοινή γεωργικής πολιτικής που θα πρέπει να εξασφαλίζει δύο και οικονομική και περιβαλλοντική όπως έλεγα με έναν τομέα ο οποίος θα αντλεί τα προς το ζήν τροποντινά, αλλά και θα έχει καλές οικονομικές επιδόσεις χρησιμοποιώντας, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους Κατά τρόπο ισορροπημένο. Πώς θα γίνει αυτό. Ε, για πολλά χρόνια ο Γεωργός είχε οφηθεί προς μια παραγωγικότητα χωρίς όρια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ευάλωτα ε, οικοσυστήματα, οι φυσικοί πόροι, πράγμα το οποίο ε, πλέον πληρώνει με διαρκείς ε, κατηγορίες ότι είναι ε, ρηπογόνα η δραστηριότητά του, ότι είναι ρηπαίνων δηλαδή ο Γεωργό. Πράγμα το οποίο όμω εμεί δεν πρέπει να επιτρέψουμε και θα πρέπει να ενισχύσουμε τον Γεωργό, να τον οθήσουμε να λαμβάνει υπόψη στοιχεία μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή του, χρησιμοποιώντας δηλαδή πρακτικές παραγωγής βιώσιμες αηφόρες. Αυτές υπάρχουν, μπορούμε να τις βελτιώσουμε ακόμη όλοι μαζί και στόχο έχουν να εξασφαλίσουν το στόχο της ε, διατροφικής ασφάλειας μακροπρόθεσμα. Μπορεί δηλαδή ένα ξέφατο στο δάσος να διαφυλάσει από τη διάβρωση το έδαφος. Ε, δεν σημαίνει ότι είναι έδαφος χαμένο από την παραγωγικότητα, από τη γεωργική παραγωγή. Όχι, γιατί αυτό ε, αυτό το ξέφωτο επιτρέπει την διάσωση ολόκληρη τη περιοχή, την αηφορία δηλαδή τη παραγωγή σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό πρέπει να το καταγράψουμε στα θετικά στοιχεία τη ε, παραγωγή και γι' αυτό προτείνουμε να σα ε, δώσουμε σαν ιδέα τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, την διαφύλαξη των βοσκοτόπων, την προστασία του περιβάλλοντος. Επιλογές ω προ έναν αριθμό περιορισμένων μέτρων που θα εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί επιτρέπουν αυτά τα μέτρα και να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, η απώλεια δηλαδή βιοπικιλότητα, η διάβρωση των εδαφών αντιμετωπίζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό και απλό. Ταυτόχρονα όμω ούτε ο γεωργό ούτε και η γραφειοκρατία επιβαρύνονται υπερβολικά με ε, δυσβάσταχτα μέτρα. Πρόκειται για μέτρα τα οποία είναι εφαρμόσιμα σε ολόκληρη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι μπορεί ο Γεωργός με τον τρόπο αυτόν να στηριχθεί γιατί προτείνονται τα ίδια μέτρα για όλους τους Γεωργούς είτε ε, και, μπορούν να εφαρμοστούν από τη Φιλανδία μέχρι την Ισπανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την ε, Πολωνία. Με το μηχανισμό αυτό θεωρούμε ότι και οι γεωργοί και οι φορολογούμενοι είναι σε μια θέση που σίγουρα θα κερδίσουν. Μετά θα, θα καταβάλουμε μια προσπάθεια για την γεωργία της γνώσης. Παράλληλα, θα αναπτύξουμε νέα μέσα για την έρευνα και την καινοτομία. Η γεωργία του αύριο είναι η γεωργία της γνώσης. Είναι η υλοποίηση στην πρακτικά αυτή της έννοιας που θα μας επιτρέψει να παράγουμε περισσότερα με λιγότερα μέσα. Να συμφιλιώσουμε τις οικονομικές και οικολογικές πτυχές και να προωθήσουμε το γεωργικό τομέα και σε περισσότερη ανταγωνιστικότητα και σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα και με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μια καλύτερη προσαρμογή στην ζήτηση ε, και στις, ε, θα συνδυάσουμε τη ζήτηση και τις, ε, τους περιορισμούς τη παραγωγή. Γι' αυτό προτείνω στις δημοσιονομικέ προοπτικές να διπλασιάσουμε την προσπάθεια όσον αφορά τη γεωργική έρευνα. Δεν χρειάζεται να χρηματοδοτήσουμε μόνο τι εργασίε του εργαστηρίου, διότι εάν έστω και αν είναι οι καλύτερες ιδέες αυτές που βγαίνουν από το εργαστήριο, εάν δεν εφαρμοστούν είναι άχρηστες. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τεχνολογίες που να ε, ε, χρειάζονται στους γεωργούς, θα πρέπει να διευκολύνουμε τις μεταφορές γνώσης, να ε, ενισχύσουμε τις σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στην γεωργική κοινότητα και στην επιστημονική κοινότητα. Αυτοί οι στόχοι κλειδιά θα μπορούσαν να θέσουν τις βάσεις μιας πραγματικής ε, γεωργίας της γνώσης και θα αποτελέσουν τον πυρήνα μιας συνεργασίας για την καινοτομία που θα επιτρέψει να κινητοποιήσουμε όλα τα κοιτάσματα αν θέλετε παραγωγικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα... Και, αυτά, και οι προτάσεις, θα υποβάλουμε προτάσεις για το θέμα αυτό στο άμεσο μέλλον που θα έχουν άμεση σχέση με τις προτάσεις που κάνουμε σήμερα. Τώρα, ε, θα οργανώσουμε τους διάφορους κλάδους ε, έτσι ώστε να υπάρχει μια βιώσιμη κατανομή της προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα με την ε, οικολογική βιωσιμότητα, την καινοτομία και την έρευνα θα πρέπει να έχουμε τα επόμενα χρόνια εργαλεία οικονομικής βιωσιμότητας. Στο εσωτερικό της διατροφικής αλυσίδας όπου ο πιο σημαντικός κρίκος είναι η πρωτογενής γεωργική παραγωγή και που είναι και ο πιο ευάλωτος, θα πρέπει να ε, επαναφέρουμε την ισορροπία και να ενισχύσουμε την θέση των ε, γεωργών. Θα πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη κατανομή τη ε, προστιθέμενης αξία. Γι' αυτό προτείνω να δώσουμε την δυνατότητα σε όλου του γεωργού, ε, όπω προβλέπεται στου τομεί που καλύπτονται από το παράδειγμα 1 τη συνθήκη, να οργανωθούν. Δεν κοστίζει τίποτα και είναι μια προσφορά, δηλαδή προσφέρουμε ένα νομικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στι ανάγκε του, των γεωργικών δραστηριοτήτων, των κλάδων της βιομηχανίας, που μπορεί να προσφέρει όμως πολλά στους, γεωργικούς, στους παραγωγούς για να μπορέσουν να τοποθετηθούν πιο αποτελεσματικά στην αγορά. Πιστεύουμε ότι οι αγορές αυτές, οι οργανώσεις μάλλον αυτές, ε, θα βοηθήσουν τους γεωργού και είναι ανοιχτέ σε όλου του τομεί. Επίση, όταν οι επαγγελματίε θα το ζητήσουν, προτείνουμε την αναγνώριση από πλευράς των κρατών μελών των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων των οργανώσεων των παραγωγών και των διαπαγγελματικών οργανώσεων και η αναγνώριση αυτή πρέπει να είναι υποχρεωτική. Προτείνω να διευκρινίσουμε τους κανόνες ανταγωνισμού. Τίποτα δεν δικαιολογεί να εμποδίσουμε την οργάνωση των παραγωγών, να διασφαλίσει ε, μια, μια οργάνωση αν θέλετε, ε, μια προσαρμογή της παραγωγής στην, ε, στη ζήτηση της αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Αυτή η οργάνωση θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια οικονομική ε, βιωσιμότητα παράλληλα με τα άλλα εργαλεία τα οποία σας είπα και θα επιτρέψει στους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τις διάφορες κρίσεις. Τώρα, ποια είναι τα ε, σύγχρονα όργανα διαχείρισης των κρίσεων. Προτείνουμε μια, ένα απόθεμα κρίσης 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για τα μέτρα στην αγορά σε περίπτωση κρίσης ε, στην αγορά ή απώλειας εμπιστοσύνης από πλευράς ε, των καταναλωτών σε μεγάλη κλίμακα. Επίσης προτείνουμε μια ρήτρα ε, έκτακτης ε, διακύμανσης ή διαταραχής, ε, κρίσης για να καλύψουμε τα, τα, τις απρόβλεπτες ε, κρίσεις, τα απρόβλεπτα προβλήματα. Θυμόσαστε τι έγινε με την κρίση με το e-call τελευταία ή τις διάφορες ε, υγειονομικές ε, κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας. Θα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι να μπορέσουμε να, αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τα προβλήματα άμεσα. θα πρέπει, η παρέμβαση ή η ιδιωτική αποθεματοποίηση λειτουργική όμως ε, η έκτακτα συμπληρωματικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα. Θα πρέπει να, δράσουμε άμεσα χωρίς να περιμένουμε να ε, διονγκωθεί η κρίση, χωρίς να περιμένουμε να ε, γονατίσει πραγματικά ο γεωργικός ε, τομέας. Δηλαδή θέλουμε να, είμαστε, να αντιδρούμε άμεσα και να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτά είναι, αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά. Τώρα, μέσα στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, ένα νέο εργαλείο διαχείρισης των κρίσεων, το εργαλείο καταπολέμησης της των άμεστων των αλλαγών ε, που θα έχει σαν φιλοσοφία βοήθησε τον εαυτό σου και η Ευρώπη θα σε βοηθήσει. Δηλαδή, κάνετε κάποιες ασφάλειες, ε, ασφαλιστείτε, δημιουργήστε κάποια ταμεία και η Κομισιόν θα σας βοηθήσει, θα σας υποστηρίξει. Τώρα, εδαφική διάσταση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας στο σύνολο των, ευρωπαϊκών εδαφών. Δεν θα, θα πρέπει να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό των εδαφών. Θα πρέπει να υποστηρίξει η ΚΑΠ την εδαφική συνέχεια της γεωργίας. Θα πρέπει να έχουμε μια διακυβέρνηση πιο αποτελεσματική που θα εστιάζεται σε συγκεκριμένους στόχους και αυτό προτείνουμε εμείς η Κομισιόν προτείνει στα κράτη-μέλη να προχωρήσουμε προς μια νέα διακυβέρνηση η οποία θα στηρίζεται σε συμφωνίες συνεργασίες ανάμεσα στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη όπου θα συμπεριλαμβάνονται τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Η προσέγγιση του, ε, της Σύμβασης ε, Συνεργασίας θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ και άλλων μηχανισμών εθνικού συντονισμού και με, με την Κομισιόν ε, κάποιους, ε, εξάντε που θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί από τα κράτη-μέλη πριν την έγκριση των προγραμμάτων αυτών από την Κομισιόν. Θα επιτρέψει επίσης την διευκόλυνση εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι οι κοινοί κανόνες ε, ανάμεσα στην ανάπτυξη της υπαίθρου και τα διευθυντικά ταμεία θα οδηγήσουν σε κοινέ, σε γενικές αξίες και, τον, ε, και σε έναν εθνικό στρατηγικό συντονισμό και σε μια ιδιαιτερότητα της ΚΑΠ και σε, θα δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στους δύο πυλώνες. Δεσμεύομαι να συνεργαστώ ε, στενά με τα κράτη-μέλη σε αυτή την προπαρασκευαστική φάση για να περιορίσουμε τα προβλήματα, ε, τις απορίες και τις ανάγκες προσαρμογής ε, μετά την έγκριση των προγραμμάτων. Ένα καλό, μια καλή προπαρασκευαστική εργασία θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε συνεκτικές στρατηγικές σαφείς πριν από την υιοθέτηση των προγραμμάτων για να, και είμαστε σίγουροι ότι ε, θέλουμε να υπάρχει ένα συντονισμός ανάμεσα στους, στο Διδαστατικό Ταμείο και στο Ταμείο το Γεωργικής ε, και στο Γεωργικό Ταμείο της Ανάπτυξης της Υπέθρου και ταυτόχρονα όμως ε, εξασφαλίζουμε τις σχέσεις ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο πυλώνα διότι όλα ε, τα στοιχεία της ανάπτυξης της υπαίθρου παραμένουν στον κανονισμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου και συνάδουν με, το περιεχόμενο του πρώτου πυλώνα. Επομένως τα κράτη-μέλη δεν, θα είναι, ε, δεν θα συνδέονται με άξονες, μπορούν να καθορίζουν με ευέλικτο τρόπο τις στρατηγικές για την αξιολόγηση του τοπικού δυναμικού μέσα στα πλαίσια όμως των κοινοτικών στόχων αλλά η υποχρέωση εφαρμογής κάποιων μέτρων όπως ε, τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ε, ή οι προσεγγίσεις του Λίντερ θα παραμείνουν. Η διακυβέρνηση αυτή θα επιτρέψει τον εξυγχρονισμό της ε, υπαίθρου μέσω επενδύσεων στις δημόσιες υποδομές, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές υποδομές θα ενισχύσουν τον, και θα δημιουργήσουν έναν δυναμικό γεωργικό τομέα καινοτόμο που θα επιτρέψει στα εδάφη να ε, χρησιμοποιηθούν και σε μη γεωργικές ε, δραστηριότητες. Τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν ε, υποπρογράμματα περιφερειακά, εξειδικευμένα, για να βοηθήσουν στον εξυγχρονισμό των ιδιαιτέρων τομέων σε περιοχές όπου οι τομείς αυτοί παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό θα γίνει σε κάποιες, ε, σε κάποιες περιοχές, για κάποιους τομείς, ε, για να εξασφαλίσουμε μια πολυετή ανάπτυξη πιο ευέλικτα μέτρα και πιο συγκεντρωμένα για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των ζωνών της υπαίθρου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την καινοτομία, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να προωθήσουμε την, μια καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των κινδύνων, να διασφαλίσουμε τα οικοσυστήματα, να ενθαρρύνουμε την ουσιαστική χρησιμοποίηση των πόρων και να προωθήσουμε την κοινωνική συνοχή μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο προβλέπονται 20 ε, μέτρα μεταξύ αυτών. Ένα συνεκτικό πακέτο για την ε, γεωργία της γνώσης ε, με την υποστήριξη πιο συγκεκριμένα της μεταφοράς των γνώσεων, υπηρεσίες συμβουλευτικές ή ενημερωτικές, εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και ε, συνεργασία ανάμεσα στους γεωργούς και στους επιστήμονες. Μια συμπροματική προσπάθεια ε, για την ε, γεωργία η οποία στρέφεται προς την ποιότητα. Θα υπάρξει μια υποστήριξη ύψους μέχρι 3.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση για διαδικασίες που προωθούν την ποιότητα και την πιστοποίηση. Μια πραγματική στρατηγική τώρα για μια γεωργία που επενδύει, δηλαδή ενισχύουμε τις επενδύσεις στην γεωργία. Πιο αποτελεσματικά εργαλεία θα είναι διαθέσιμα για να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις στα πλαίσια ενός μέτρου όπου συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες ε, επενδύσεων με την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προσφέρουν ε, ενισχύσεις υψηλότερες για επενδύσεις ε, που δίδονται σε νέους γεωργούς, ενισχύσεις σε περιοχές, καινοτόμες επενδύσεις και συλλογικές επενδύσεις. Μία σαφής υποστήριξη σε μία οργανωμένη γεωργία που, που κυκλοφορεί τα προϊόντα καλύτερα στο εμπόριο. Θα ενισχύσουμε την, τον οργανισμό και την οργάνωση μάλλον ε, με μηχανισμούς για την ε, δημιουργία και την διατήρηση ε, ομάδων παραγωγών που θα είναι ανοιχτές στο σύνολο των κρατών μελών και τα παλιά και τα καινούρια. Η συνεργασία αυτή θα υποστηριχθεί, οι συλλογικές πρωτοβουλίες όπως παραδείγματο χάρη η δημιουργία σύντομων δικτύων θέσης εμπορία, οι συλλογικές προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, η συνεργασία ανάμεσα σε μικρούς οικονομικούς παράγοντες ε, που θέλουν να συνενωθούν θα ενισχυθούν. Οι ομάδες ε, τοπικής δράσης του Λίντερ θα ενδυναμωθούν. Μιλάμε και, για, και θα βοηθήσουμε και ε, παράγοντες που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό. Επίσης θέλουμε να υπάρξει μια νέα μια ανάπτυξη, μάλλον θέλουμε να αναπτύξουμε μια γεωργία που θα είναι πηγή απασχόλησης ε, και πνεύμα εμπορικότητας ε, και επιχειρηματικότητα συγγνώμη, στην περιοχή ε, και θα ενισχύσουμε τις μικρές εκμεταλλεύσεις και την οικονομική διαφοροποίηση, μη γεωργική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων με μια υποστήριξη η οποία θα μπορούσε να ανέλθει μέχρι το ποσό των 70.000 ευρώ. Τώρα, υπάρχει ένας εγκάρσιος στόχος που είναι η απλούστευση της ΚΑΠ. Για το σύνολο όλων αυτών των συστημάτων και των εργαλείων προτείνουμε να λάβουμε υπόψη μας μια επιτακτική εντολή που είναι η απλούστευση. Ε, είτε πρόκειται για άμεσες πληρωμές, ε, είτε ε, έχουμε, και αν έχουμε μια καταποκοπήν υποστήριξη από 500 έως 1000 ευρώ, και αυτή η ενίσχυση δεν θα εμποδίσει την αναδιάρθρωση διότι ταυτόχρονα η εκχώρηση των εδαφών από τους μικρούς παραγωγούς που σταματάνε την γεωργική τους δραστηριότητα σε άλλες ε, εκμεταλλεύσεις θα ε, ενισχυθεί μέσω ενός νέου μέτρου αναδιάρθρωσης στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα ενθαρρύνοντας την έξοδο των μικρών γεωργών ε, αν και εφόσον τον επιθυμών, το επιθυμούν. Δηλαδή θέλουμε να προβλέψουμε, προβλέπουμε μάλλον ένα μέτρο απλής, απλούστευσης των πληρωμών για τους μικρούς παραγωγούς στον πρώτο πυλώνα, αλλά δεν θέλουμε οι γεωργοί, οι μικροί γεωργοί τα να, να παραμένουν στην γεωργία για να πάρουν αυτέ, αυτές τις, ε, τις επιδοτήσεις, αυτές τις ενισχύσεις. Οι, αυτοί όμως που αποχωρούν λόγω ηλικία και τα λοιπά μπορούν να το κάνουν και θα έχουν μια ενθάρρυνση μέσω του δεύτερου πυλώνα. Τα μέτρα πρασινίσματος αν θέλετε ε, έχουν ε, προταθεί και θα ελέγχονται και θα πληρώνονται ταυτόχρονα ταυτόχρονα και μέσω των ιδίων ε, δομών όπως ε, οι βοήθειες ε, με βάση το εισόδημα. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχουν να γίνεται ταυτόχρονα ο, ο, έλεγχος, διότι δεν θέλαμε με κανέναν τρόπο να πολλαπλασιάσουμε τους ελέγχους ή την χαρτούρα και για τους γεωργούς αλλά και για τις εθνικές, την εθνική διοίκηση. Επομένως εξασφαλίζουμε μια μεθοδική διαχείριση του δημόσιου χρήματος, περιορίζουμε ταυτόχρονα το, το βάρος των ελέγχων, ε, παραδείγματος χάρη, ενισχύοντας τα κράτη-μέλη, ε, ανταμείβοντας τα κράτη-μέλη, τα οποία ε, για πολλά χρόνια ε, είχαν ένα ποσοστό λάθους κάτω από 2%. Επίσης, η ε, οι πληρωμές με βάση το, το εισόδημα, ε, ο τρόπος με τον οποίο θα χορηγούνται οι, οι, βοήθειες αυτές θα είναι πολύ πιο απλός, θα ε, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους στόχους για τους γεωργούς και για το περιβάλλον. επίσης, ο αριθμός των ΓΑΕΚ e θα περιοριστεί από 15 σε 8 και 5 απαιτήσει δηλαδή θα εξαφανιστούν. Θα λάβουμε υπόψη μας ε, επίσης στο διάφορα στοιχεία του τοπίου όσον αφορά τα δάση, τα αλσίλια, τους φράκτες κτλ. στο πλαίσιο του 7% των οικολογικών αποθεμάτων που θα πρέπει να πετύχουμε. Η γεωργία κυρίες και κύριοι είναι στον πυρήνα των τοπικών δυναμικών. Ε, πρέπει να την υποστηρίξουμε. Είναι η τροφή μας αλλά επίσης είναι και ένα ε, σύνολο ε, δημοσίων αγαθών είναι η κουλτούρα μας, είναι οι παραδόσεις μας, είναι οι αξίες μας, είναι οι δημόσιοι πόροι μας, οι φυσικοί μας πόροι, είναι το μέλλον των εδαφών μας ε, και της κληρονομιάς μας. Και τώρα ξεκινάει μια ουσιαστική φάση συζητήσεων πάνω στις προτάσεις της Κομισιόν. Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτές οι συζητήσεις θα γίνονται επίσης όρις ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Είναι μια ιστορική, ε, μια ιστορική ευκαιρία για την κοινή γεωργική πολιτική, πρέπει να υποφεληθούμε πλήρω. Ε, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε οι προτάσει ε, που υπέβαλε η Κομισιόν να με τι δικέ σα προτάσει και τι προτάσει του, του, Συμβουλίου να ε, μα οδηγήσουν σε απλά μέτρα τα οποία να μπορούν να εφαρμόσουν οι γεωργοί και να διασφαλίσουμε την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα τη γεωργία μα μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Επίτροπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ πλούσια παρουσίαση που μας έκανες. Θέλω να σας ε, διαβεβαιώσω ευθύς εξ αρχής ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να έχουμε μια συνεργατική προσέγγιση και να βρούμε με το Συμβούλιο κάθε δυνατή ευκαιρία ώστε από αυτή τη μεταρρύθμιση να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις απαραίτητες απαντήσεις στις πολυάρθμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μας. Ζητώ συγγνώμη στο ότι δεν ανέφερα κάποιες ε, παρούσες οργανώσεις, αλλά έχω ένα κατάλογο. Ευχαριστώ συνολικά όλους του παρόντες, ακόμα και αυτούς που δεν ανέφερα, όπως και τέος συναδέλφου, ε, τέος Επιτρόπου και άλλου συναδέλφου. Έχουμε πραγματικά πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί ο Επίτροπος επέλεξε να έρθει καταχάς εδώ, στο Κοινοβούλιο, προτού δηλαδή ε, δώσει σχετική συνέντευξη τύπου. Και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε κάποιο χρόνο. Και όπω σα είπα, το δεκάμιση πρέπει να αποχωρήσει. Οφείλω να σα πω όμω ευθύ εξ αρχή ότι έχουμε προγραμματίσει και μια άλλη μέρα, το συντομότερο δυνατό για να συνεχιστεί η συζήτηση που ξεκινά σήμερα. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με τον Επίτροπο για να μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητα σε όλου του συναδέλφου που θέλουν να παρέμβουν. Και τώρα ξεκινάμε με την σειρά των συντονιστών και των εισηγητών και βέβαια στη συνέχεια μετά τις πρώτες 10 παρεμβάσεις θα δώσω το λόγο και πάλι στον Επίτροπο για να δώσει κάποιες σχετικέ απαντήσεις. Είναι προφανές ότι θα δούμε καθώς θα κινούμαστε και θα πρέπει όμως να τα χειριστούμε στο το χρόνο. Ξεκινώ με τον Άλπερτ Μπέση που έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Αγαπητέ Παόλο, αξιότιμοι κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Εκ μέρους του ΕΛΚΑ θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κύριε Επίτρεπε Τσόλος και να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων και ιδιαίτερος για το γεγονός ότι ήρθατε πρώτα στο Κοινοβούλιο. Παρακολουθούν εκατομμύρια γεωργοί σε όλη την Ευρώπη με μεγάλη προσοχή τα όσα έχει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της γεωργικής πολιτικής. Και ιδιαίτερα τα μέλη της Γεωργικής Επιτροπής αναμένουν ε, με ανυπομονησία τη συζήτηση για τη γεωργική μεταρρύθμιση, τη συζήτηση αυτή που ξεκινάει σήμερα. Μέσα σε ε, αίσθημα ευθύνη το Κοινοβούλιο θα επιτελέσει το έργο του στη διαδικασία της συναπόφασης θα ήθελα λοιπόν, κύριε Επίτροπε, να έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε τις αποφάσεις μας να θα έχουμε και τα επακριβή στοιχεία για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αναφέρατε και εσείς αυτό. Ε, περιμέναμε αρκετό καιρό. Έχουμε και αρκετό χρόνο μπροστά μας, πιστεύω, για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για, την, ε, για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Κάποια στοιχεία στα οποία θα ήθελα να, επισέλθω, είναι το 30% των άμεσων πληρωμών, το 7% της οικολογικής αγρανάπαυσης, το 10% για τους ε, ε, περιστασιακούς γεωργούς και το 10% ε, επίσης για τους νέους γεωργούς είναι ζητήματα στα οποία θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση έτσι ώστε να καταστεί ανταγωνιστική η γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι με την ε, συζήτηση θα βρούμε ε, το σωστό δρόμο τις σωστές λύσεις έτσι ώστε να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Γεωργία σε όλες τις διαφορές. Χρειάζεται δηλαδή ευελιξία στα μέτρα και θεματικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά διαφορετικά που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά Φιλανδία και Σικελία. Ε, δεν θα μπορούσε να έχουμε μεγαλύτερε διαφορέ στην ε, διαμόρφωση του γεωργικού ορίζοντα από τη μια άκρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην άλλη. Και γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει επουδενή τα μέτρα που θα εισαχθούν να επιφέρουν ε, ε, επιπλέον γραφειοκρατικό βάρος, το οποίο αναφέρατε και εσείς, ως πρόθεση, αν και εγώ ανησυχώ για αυτό το ενδεχόμενο Επίση, υποχρεωτική αγρανάπαυση θα πρέπει να αποφευχθεί γιατί μπορεί να οδηγηθούμε σε πολύ ψηλότερε τιμέ ε, στα προϊόντα. Ε, μέτρα περιβαλλοντικά που υφίστανται αυτή τη στιγμή και συνεχίζει η λειτουργία τους δεν θα πρέπει να ε, τεθούν σε δυσμενέτερη θέση γιατί έχουν αποδείξει την το όφελός τους στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και το περιβάλλον. Η εισαγωγή των νέων μέτρων δεν θα πρέπει να ισοδυναμεί με ε, κυρώσεις για τον Γεωργό, δηλαδή με περισσότερη γραφειοκρατία. Θετικό βλέπω ως, ιδιαίτερο ε, ιδιαίτερο θετικό στοιχείο βλέπω ότι ε, μιλάτε για την καινοτομία, για την ενίσχυση των γεωργών. Αναγνωρίστε τον ρόλο κλειδί που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Γεωργία και κυρίως μέσα στις νέες προκλήσεις της εποχής. Στο δεύτερο πυλώνα λοιπόν θα θέλαμε περισσότερη ευελιξία και συμφωνώ μαζί σας ότι έχουν ξεπεραστεί οι παλαιές δομές, πρέπει να βρούμε νέες δομές με σωστή προσθέμενη αξία και φυσικά σε αυτό θα συμβάλλει το Κοινοβούλιο όσο μπορεί. Κύριε Επίτροπε, ελπίζω ότι στις διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα που κι εσείς εξαγγέλλετε Ελπίζω λοιπόν ότι σε αυτές τις πραγματεύσεις θα συνεργαστείτε στενά με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να βρούμε μαζί καλές λύσεις. Το Κοινοβούλιο ιδιαίτερα θα πιέσει στην εξέβρεση, στο στόχο της εξέβρεσης των λύσεων που θα δώσουν τις σωστές απαντήσεις εναντί των μεγάλων προκλήσεων του μέλλοντος. Απαντήσεις οι οποίες θα ωφελήσουν τη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε να μεριμνήσουμε για την διατροφική ασφάλεια, για την υψηλιστική ασφάλεια 500 εκατομμυρίων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το μέλλον. Να μπορεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον να εξασφαλίζει επαρκή τρόφιμα για τον πληθυσμό της. Αυτό είναι ο κύριος στόχος, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και πιστεύω ότι στο προσεχές διάστημα με καλή συνεργασία θα μπορέσουμε να τον επιτύχουμε. Εύχομαι σε όλους μας καλή επιτυχία για το καλό του Ευρωπαίου Γεωργού. Να βρούμε καλές λύσεις δηλαδή. Είναι μια καλή βάση για συζήτηση οι προτάσει σα τι ε, θετικέ εξ αυτών θα τι υποστηρίξουμε. Εκεί όπου βλέπουμε ότι χρειάζονται κάποιε αλλαγέ, βεβαίω θα καταθέσουμε τι σχετικέ προτάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Άλμπερτ. Και τώρα δίνω το λόγο στον Λουίς Κάπλα Σαντόσο, συντονιστή, αλλά και εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Κύριε κύριοι, καταρχάς. Καλωσορίζω το γεγονός και το χαιρετίζω το ότι ήρθατε καταρχάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξηγήσετε και να παρουσιάσετε τις νέες προτάσεις για την ε, νέα ΚΑΠ. Και αυτό βέβαια υπογραμμίζει τις πολύ καλές σχέσεις που ήδη έχετε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ΚΑΠ είναι προφανώς μείζον πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αποφάσεις οι οποίες πρόκειται να ληφθούν θα είναι εξαιρετική σημασίας και είναι εξαιρετικά σημαντικό και στα πλαίσια της συνθήκη Λισαβόνας. Πρέπει λοιπόν να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να συνεισφέρουμε στην λήψη μιας απόφασης για μια Ευρώπη πολύ πιο ισχυρή και για την επανάκτηση των αξιών αλληλεγγύης και δικαιοσύνης που ήταν και η βάση του όλου ευρωπαϊκού ιδεώδους οικοδομήματος. Ως εισηγητής των σοσιαλιστών θα είμαι πιστός στην απόφαση που ελήφθη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του θέματος. Θα είμαστε όμως και επαρκώς ευέλικτοι και διατηθέμενοι σε διάλογο με τους συναδέλφους πολιτικές ομάδες στις όλες διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και με την Επιτροπή στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας ικανοποιητικής ανταπόκρισης και ισόρροπης απάντησης. Η ομάδα των σοσιαλιστών είναι σαφέ ε, ότι βέβαια έχω κάποιο ρόλο συντονιστού, αλλά βέβαια έχουν απόλυτη επίγνωση του ρόλου και τη ευθύνη του. Πρέπει να αναλάβουμε στα πλαίσια των διαδικασιών για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ, θα πρέπει με συνοχή και με συνενετικό και συμβιβαστικό πνεύμα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Επαναβεβαιώνω λοιπόν τη βούλησή μα να συνεισφέρουμε στο τελικό αποτέλεσμα που θα ανταποκρίνεται στι ευχέ όχι μόνο των καταναλωτών, αλλά εν γέννη των Ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών σε ό,τι αφορά την ε, ουσία της μεταρρύθμισης, οφείλω να πω ότι σε σχέση με τους στόχους ε, των υποθέσεων εργασίας και αρχιτεκτονικής υπάρχουν πολλά θετικά ζητήματα, αλλά γύρονται πολλές ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ε, πρακτική εφαρμογή όλων, όλης αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, που είναι και το πλέον σημαντικό βέβαια. Προτού εκφραστώ σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη αυτή πρόταση και μπορώ παρουσιάσω συγκεκριμένες θέσεις, οφείλω να, να εξηγήσω πού έγκυται η διαφωνία μου με το μέγεθος ε, και το μερίδιο του ΑΕΠ, του κοινοτικού Προϋπολογισμού που δίνεται στην ΚΑΠ. Αυτή δεν είναι... Ε, ήδη στο παρελθόν έχουμε εκφράσει με συντριπτική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποια θα έπρεπε να είναι το επαρκές, ε, επαρκής προϋπολογισμός για μια ΚΑΠ. Η ΚΑΠ δεν μπορεί να καλύψει τους ε, στόχους της χωρίς επαρκή προπολογισμό με το τέλος του 2014 ολοκληρώνεται η φάση phasing in για τα τελευταία κράτη-μέλη και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ισότιμα από το 2000, ε, τέλος 2014 και επέκεινα. Ως εκ τούτου λοιπόν πιστεύω ότι είμαστε, λίγο, είμαστε ε, πολύ πιο κάτω από τις ε, προσδοκίες μας. Σε κάποιους τομείς είναι πολύ δηλές οι προσπάθειες, σε άλλες είναι πραγματικά παράδεκτες. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ανακατανομής και της σύγκλησης των άμεσων πληρωμών μεταξύ γεωργών και κρατών μελών. Η πρόταση ως έχει, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πραγματικά η ελάχιστη κακατούρα των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί. Για παράδειγμα, στην ε, Λετωνία υπάρχει μια μείωση των άμεσων πληρωμών όπου θα λαμβάνουν λιγότερο από το 50% των άμεσων πληρωμών. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το 2020 ουσιαστικά η χώρα αυτή θα λάβει μόλις το 60% του ισχύοντος, του τρέχοντος μέσου όρου της ε, κοινότητας. Και αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός ε, σύγκλησης και πριν από το 2040 η Λετωνία θα φτάσει το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η όλη καθάση λοιπόν θεμελιώδης. Εμείς οι σοσιαλιστές είμαστε κατά βάση και κατ' ουσίαν σύμφωνοι με τους περιβαλλοντικά κριτήρια και την αντιστάθμιση παραγωγής ε, δημοσίων ε, ωφελιών από τους ε, γεωργούς που είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας. Ως εκ τούτου λοιπόν όντως αξίζουν και πρέπει οι γεωργοί να έχουν και άμεσες πληρωμές. Είναι λοιπόν απαραίτητο όχι μόνο να καθορίσουμε αντικειμενικό τρόπο επί τη βάση υπολογισμού την αποδεκτή επιφάνεια κάθε κράτο μέλο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει σε κάθε υπολογισμό απόλυτα αντικειμενικό τρόπο και ελάχιστα γραφειοκρατικό για να υπάρχει πρόσβαση σε αυτέ τι άμεσε πληρωμέ. Έχω σημειώσει την προσπάθεια που σκοπεύει να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Η ομάδα μου είναι πρόθυμη να παρουσιάσει σχετικέ προτάσει. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ενεργού γεωργού, που είναι μια νέα έννοια και την οποία είμαστε πολύ ευνοϊκά διακείμενοι, πέρα από το γεγονότος βέβαια, παρά το γεγονός ότι η δική σας πρόταση η, ο, ορισμός που δίνεται είναι καλύτερος από τις φήμες που ακούγαμε τελευταία, εν θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ παραπάνω πάνω σε αυτή την πρόταση αυτή. Ένας αγρότης δηλαδή ο οποίος μπορεί να δέχεται μια δημόσια χρηματοδότηση, ένας αγρότης ο οποίος ε, λαμβάνει τέτοια δημόσια χρηματοδότηση, θα πρέπει να ξέρουμε και ποιο είναι το ποσοστό του εισοδήματός του που προέρχεται από την, αμυγή γεωργική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής η Βασίλισσα της Αγγλίας εξακολουθεί να είναι ενεργός, ε, ενεργή στη Γεωργία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και να γίνεται αποδεκτό στη νέα ΚΑΠ και να βαρύνει τον φορολογούμενο. Και ας περάσουμε στο δεύτερο πυλώνα. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα ο αποκλεισμό ε, της ενίσχυσης ε, στις επενδύσεις. Σε επενδύσει σε νέους τομείς. Ε, πώς είναι δυνατόν να αποκλείεται η υποστήριξη στις ε, στα νέα αρδευτικά έργα που είναι ένα από τα μέσα για να μπορέσει να καταπολεμηθεί η απερίμωση ε, και η απερίμωση η οποία παρατηρείται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Χωρίς νέα αρδευτικά έργα δεν είναι δυνατόν να είναι ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αυτή η παράληψη λοιπόν θα πρέπει να καλυφθεί κύριε Επίτροπε και θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό της αγοράς που είναι επίση θεμελιώδης όπως είπε και ο Επίτροπος σε εποχές εξαιρετικής μεταβλητότητας των τιμών και αστάθειας των αγορών ε, παρά τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ε, η πρόταση θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δειλή και άτολμη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κανονισμό των νέων χρηματοδοτικών μέσων. Ω εκ τούτου θα μιλήσουμε για τα σχετικά πλέον εκτήματα και μειονεκτήματα όταν θα έχουμε μελετήσει ει βάθο και λεπτομέρω την πρόταση αυτή. Δεν μπορώ ε, να. Ε, μακρηγορήσω σε αυτό, αλλά να, να κάνω κάποια σχετικά σχόλια ακόμα. Αναγνωρίζουμε ότι είναι καλό εφαλτήριο η πρόταση αυτή και είμαστε διατεθειμένοι να διευκολύνουμε, να βελτιώσουμε κάποιες προτάσεις, όπως για παράδειγμα το ειδικό καθεστώς των ε, γεωργών, ε, το ζήτημα της ε, δυτής ε, εκμετάλλευσης των νεαρών γεωργών που είναι πολυθετικό όπως και η ενίσχυση των επαγγελματικών οργανώσεων των παραγωγών, των διεπαγγελματικών οργανώσεων, τις εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για την καινοτομία και την έρευνα, καθώς και μια μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών ταμείων. Ολοκληρώνω, κύριε Επίτροπε, επαναλαμβάνοντα αυτό που γνωρίζουμε οι πάντε, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, εξαιρετικά βέβαια προκλητικό και ε, ενδιαφέρον, και το οποίο όλοι έχουμε μεγάλο ενθουσιασμό να συνεργαστούμε στενά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ξεβρεθεί μια λύση που θα είναι ικανοποιητική για την Ευρώπη, για του Ευρωπαίου γεωργού και πολίτε. Ας, προσπαθήσουμε, προχωρήσουμε όσο να πιο γρήγορα. Ο Τζόρτζ και μετά ο Νίκος. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, ξέρω ότι ε, θέλουμε να μιλήσουμε στον περισσότερο συνάδελφοι, θα είμαι σύντομος. Αυτό το πακέτο, βλέποντας το αρχικά, έχει κάποια καλά και κάποια κακά στοιχεία όσον αφορά την ε, ομάδα μας ε, το Άλτε. Αν ξεκινήσουμε με τα καλά. Μου αρέσει, καλά το, μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι στοχεύουμε καλύτερα τις πληρωμές. Καλωσορίζω την μετακίνηση ε, από την στάση που είχαμε στο παρελθόν ε, σε αυτό το οποίο λέμε τώρα, να, οι, οι ενισχύσεις να δίδονται σε αυτούς που πρέπει να δοθούν. Επίσης, ε, καλωσορίζω την ευελιξία η οποία εισάγεται και επίσης ε, καλωσορίζω και την απλούστευση της ΚΑΠΑ. Βέβαια δεν ξέρω πόσο απλή θα είναι όταν ε, αρχίσουμε και μελετάμε με λεπτομέρειες ε, τα μέτρα αυτά. Αλλά τέλος πάντων. Επίσης είναι πιο δίκαιο το σύστημα πληρωμών ανάμεσα στα κράτη και στους γεωργούς. Βέβαια είναι μικρό το βήμα και κάποιοι ίσως απογοητευτούν και θα θέλουν να κάνουμε κάτι παραπάνω. Τώρα για το ουσιαστικό θέμα το οποίο το συζητήσαμε επί μακρόν, ε, στην Επιτροπή μας και με εσάς βέβαια πάρα πολλές φορές ε, τις μεγάλες αλλαγές ε, ε, που αντιμετωπίζουμε λόγω της έλλειψης ε, εδαφών, νερού κτλ εγώ θεωρούσα και ήλπιζα ότι το πακέτο αυτό θα είχε ε, κίνητρα, θα πρότεινε κίνητρα για την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου γεωργίας που θα είναι πιο ανταγωνιστικό, ε, που θα είναι πιο αποτελεσματικό, που δεν θα παράγει τόσο πολύ ε, διοξίδιο του άνθρακα. Όμως δυστυχώς το πακέτο αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν υπολείπεται πολύ των προσδοκιών μας, δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλουμε. Για το 7% set aside ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι τελικά η γεωργία της κοινότητας κινδυνεύει να είναι λιγότερο ανταγωνιστική και όχι περισσότερο ανταγωνιστική. Η... Μιλάμε για διατροφική ασφάλεια, για ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό το 7% ε, του set aside δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Ίσως θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε, δεν ξέρω. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθεί η κοινή γεωργική πολιτική τα τελευταία δέκα χρόνια, ίσως ε, να μην, έχουμε, να μην διακόπτουμε εδώ τώρα την πορεία μας, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι κάνουμε μια μεγάλη παράκαμψη από την πορεία μας και ελπίζω να μην καταλήξουμε σε αδιέξοδο. Οι διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν θα ε, είναι μεγάλες ε, και δύσκολες και ελπίζω ότι με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου θα επαναφέρουμε το όχημα πίσω στην πορεία του. Ο Τζιμ Νίκολσον και μετά ο Μάρτιν Όσλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε εδώ. Είναι δύσκολο, όπω αντιλαμβάνεστε και εσεί ε, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να δώσουμε ανάλυση επί τη ουσία και ει βάθο των προτάσεών σα, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να δώσουμε μια πρώτη απάντηση για την κατάσταση, για τι θέσει μα και νομίζω ότι καθίσατε σαφέ στη θέση μα έστω ε, και σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ, Πρόεδρε, Έχω χρόνια σε αυτήν την επιτροπή. Έχω περάσει από, επιτρο... από μεταρρύθμιση Μαξάρη, από Φίσλερ, από μικρή μεταρρύθμιση, από μεγάλη μεταρρύθμιση Φίσλερ. Και ήταν ξεκάθαρη η κατεύθυνση που ακολουθούσε αυτή η μεταρρύθμιση. Θα ήθελα δυστυχώς να διαπιστώσω ότι είναι περίπλοκη, γραφειοκρατική η μεταρρύθμιση αυτή. Θα επιβάλλει περισσότερο δηλαδή γραφειοκρατικό άχθος στον Γεωργό και θα είναι πιο δύσκολη να τη διαχειριστεί ο Γεωργός πολύ ευχαριστώ να συνεργαστώ μαζί σα για να βελτιωθεί αυτό το χαρακτηριστικό και ελπίζω ότι και εσείς θα ανταποκριθείτε θετικά όπω και εμεί δείχνουμε διάθεση συνεργασία απέναντί σα. Γιατί όπω έχει τώρα αυτό το σύνολο των προτάσεων σα οδηγεί στην αποδιάρθρωση τη ασφάλεια τη επιστημικής αλυσίδα που χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμα για να τρέφουμε του πολίτε τη Ευρώπη. Και στον κύριο Κάπουλα Σάντο, θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι Μπορεί να αναφέρεστε στην ε, πατρίδα τη ε, μεγαλειοτάτη Βασίλισσα τη Αγγλία, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλοί γεωργοί που τη σκάβουν αυτή τη γη και τη δουλεύουν. Και θα ήθελα να δείχνετε πιο πολύ σεβασμό στην υψηλότητά τη. Περιμένω να ακούσω, αλλά αν οι διερμηνεί ε, τα βγάλανε πέρα, λέει ο κύριο ομιλητή. Η δική μου λοιπόν θέση δεν έχει αλλάξει. Και σε σχέση και με το προηγούμενο, ε, Επίτροπο. Το έχω πει ξεκάθαρα αυτό. Τα μέτρα, τα πράσινα μέτρα στον δεύτερο πυλώνα επαρκούν. Πιστεύω ότι το να τα μεταφέρουμε στον πρώτο πυλώνα απλώ περιπλέκει την κατάσταση, επιβάλλει την γραφειοκρατία. Ίσως κάποιοι να το προτιμούν. Δηλαδή θα είναι πιο, λοιπόν, πιο δύσκολο να διαχειριστεί κανείς αυτά τα μέτρα. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πούμε, ότι πρέπει αυτά τα μέτρα να τα εφαρμόσουν οι γεωργοί στα 27 κράτη-μέλη να φτάσουμε δηλαδή τη στιγμή που ο Γεωργός θα πρέπει να υλοποιήσει αυτή την πολιτική εφαρμογή και αυτό, εκτελεστική πολιτική, αυτό δεν θα είναι δυνατόν, δεν θα λειτουργήσει σωστά. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον οπισθοδρόμηση και το 7% της αγρανάπαυσης. Όταν έχουμε υψηλό κόστος των ε, σπόρων που εισάγουμε για την ε, ζωοτροφή των ζώων μας, είναι η οπισθοδρόμηση να μιλάτε για 7% τη γραμμάπαυση. Κοιτάξτε τι έχετε, και αυτό είναι ένα ασφαλό που την επέξω στο παρελθόν. Ρίξτε μια ματιά στη ζάχαρη. Έχετε αποδιαρθρώσει, έχετε διαλύσει την ε, παραγωγή σακχάριου σε όλη την Ευρώπη. Στη Ιρλανδοί έχουν βρεθεί στην ανεργία. Αυτό δεν σα έχει διδάξει αρκετά. Α μάθουμε τουλάχιστον από τα λάθη μα, α μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον. Και επίση θα ήθελα να σημειώσω Χαίρομαι για τα μέτρα στήριξη που προτείνεται σε ορισμένου τομεί και κυρίω την ταχύτερη ανταπόκριση σε περίπτωση κρίσεω. Αυτό βεβαίω το θεωρώ ευπρόσδεκτο, όπω και τα όσα είπατε για, τους, ε, για τι μικρότερε εκμεταλλεύσει θα ήθελα περισσότερο να ε, έχω πληροφορίες ότι σημαίνει ενεργός ή δραστήριος ανάλογα με το κράτος μέλος. Γιατί θα ήθελα να σας περιθυμίσω ότι σε κάθε κράτος μέλος αυτό σημαίνει κάτι διαφορετικό και δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι λοιπόν και επίσης για το επίπεδο, για το κάπινγκ θα αντιταχθώ ασφαλώς διότι ορισμένα από τα νέα κράτη-μέλη θα έχουν σαν συνέπεια μια απόλυτη καταστροφή αν εισαχθεί αυτό το μέτρο, όπως και σε ορισμένε από τι παλαιότερες περιοχές. Πρέπει να βρούμε δηλαδή λύση η οποία δεν θα παρεμποδίσει τη λειτουργία της, ε, του, την εργασία του Γεωργού, να μπορεί να κάνει ο Γεωργός την δουλειά πρέπει. Και επίση σε κάποιε περιφέρειε μικρότερε όπω η δική μου που, είναι, έχει ένα μικρό ε, αρρώσιμο τομέα. Τι θα, με, τι θα επιβάλλουν τα μέτρα αυτά περισσότερο από ότι απλώς περισσότερη γραφειοκρατία και επιβάρυνση για τον Γεωργό. Τι θα προσφέρουν περισσότερο. Γιατί νομίζω ότι εδώ έχετε κάνει λάθος. Προσπαθώντας δηλαδή να εισαγάγετε ε, ένα μέτρο τύπου unisex ε, το οποίο θα επιβάλλεται στους πάντες χωρίς ε, διαφοροποίηση έχετε αποτύχει και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον για τι ανταλλαγέ, ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ριζική μεταρρύθμιση, στη, ε, τροποποίηση μάλλον στι προτάσει αυτές και ελπίζω να υπάρχουν αρκετές παρεμβάσει συμβολές στη, συζήτηση και τροπολογίες στη συνέχεια για να τροποποιηθούν οι προτάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Μάρτιν Όσλινγκ και μετά Φοντάνο. Ναι, Πρόεδρε ανοίξατε προς την ορθή κατεύθυνση, πιστεύω, λίγο τη θύρα προς την διάσωση κοινή ελληνική πολιτική, πολιτικής, αλλά δεν αρκεί αυτό. Αν θέλουμε δηλαδή με σοβαρότητα να προχωρήσουμε σε αηφορία, σε πράσινη γεωργική πολιτική, τότε θα πρέπει να ε, προτείνουμε κάποιες σημαντικές επικρίσεις σε κάποια από τα μέτρα σας για το πρασίνισμα το λεγόμενο και το 70% το οποίο προτείνεται δεν αρκεί. Το 7% ε, επίσης ε, δεν σημαίνει ε, αγρανάπευση ουσιαστική, σημαίνει απλώς διακοπή της αξιολόγησης, της αξιοποίησης της γης. Δεν είναι πραγματική αγρανάπαυση που θα επέτρεπε να επιβιώσει το έδαφος στο πρασίνισμα. Ναι, πολύ καλά αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε σημείο αναφορά στο 2014 γιατί θα έχουμε χάσει πολύ από την πράσινη γεωργία μέχρι τότε. Και αυτό κύριε Επίτροπε που είδα και από την πρώτη έκθεσή σας γιατί δεν αναπτύσσεται μια πολιτική ευρωπαϊκή η οποία θα επιτρέπει μια ουσιαστική ε, προστασία των γεών με την αμύψη φορά. Επίσης πιστεύω ότι ο σχετισμός προς τις ε, θέσεις εργασίας έχει βρει έχει αποτελέσει μια σωστή πολιτική. Είναι κάτι το οποίο έχει στήσει το Κοινοβούλιο με ευρύτατη πλειοψηφία, αν έχουμε ανώτατα επίπεδα. Ωστόσο, δεν δίνεται τόσο θετική η λύση που έχετε βρει ως προς την ανακατανομή σε όλη την Ένωση αλλά και ιδιαίτερα ως προς ορισμένα κράτη-μέλη και δει τα καινούρια τα οποία πιστεύω θα πρέπει να συζητήσουν τα μέτρα πολύ πιο λεπτομερώς. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει θα είναι η εξοικονόμηση των τροφίμων των πόρων μας αυτών των διατροφικών διότι ξέρουμε ότι 30% τουλάχιστον των τροφίμων πάνε στα σκουπίδια. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να εξοικονομήσουμε από αυτούς τους διατροφικούς πόρους, όχι μόνο να παράγουμε περισσότερο. Και βεβαίω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα μέτρα ή ε, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε διάφορες περιοχέ τη Ευρώπη στη συνέχεια ε, στο δίλημα μεταξύ εντατικοποίησης και ε, βιώσιμης παραγωγής στη γεωργία είναι ξεκάθαρο η επιλογή θα πρέπει να κάνουμε αλλά πρέπει να ορίσουμε και σαφώς τους όρους της. Στην ε, εμπορευματοποίηση, στη διάθεση των προϊόντων πρέπει να έχουμε καλύτερα μέτρα δεν είμαι διατεθειμένο βεβαίω ε, τα χρήματα που θα διθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθώ να καταλήγουν στι ασφαλιστικέ ε, επιχειρήσει, στου ασφαλιστικού ομίλου, οι οποίοι τα ασφαλίζουν το γεωργό από την απώλεια εισοδήματο. Για δε το γάλα, βεβαίω μπορούμε να ακολουθήσουμε, αλλά εφόσον τα μέτρα είναι σωστά και αποτελεσματικά. Πρέπει να τα συζητήσουμε περισσότερο. Για το δεύτερο πυλώνα, Είναι πάλι ένα από τα πάγια αιτήματα των, των πρασίνων δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ακόμη και αν χαθεί ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ των πυλώνων ότι πρέπει να έχουμε τα πράσινα μέτρα του Λίντερ, τα πράσινα μέτρα για το Γεωργό που θα υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να διαθέτουν συγκεκριμένο ποσοστό για τα μέτρα αυτά ε, τα πράσινα ε, και δεν θα τους επιτρέπει, δεν θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη δηλαδή όλα τα κονδύλια να τα αφιερώνουν στον ανταγωνισμό και την παραγωγικότητα. Κάτι ακόμη μια και είναι πολλοί οι συνάδελφοι που μιλούν για το Γεωργό ως στοιχείο, ως παράγοντα στη γεωργική πολιτική. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτό το στοιχείο φυσικά υπάρχει. Η σημασία του, του παραγωγού, του γεωργού είναι πάρα πολύ μεγάλη για την αηφορία, για την πράσινη γεωργία. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και το ρόλο που διαδραματίζει ο καταναλωτής με τις επιλογές του στην πράσινη ε, γεωργία. Άρα πρέπει και μέσα από το πρίσμα αυτό να δούμε τα μέτρα που θα ε, εισαχθούν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ορισμένοι, ορισμένα τα οποία δεν έχουν πραγματικά επιλέξει τον δρόμο της διάσωσης της γεωργίας μας αλλά ε, κοιτάζοντας μόνο πόσα λεφτά θα μπουν στο δικό τους κορβανά, ε, παρεμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων, περιμένοντας ότι απλώς θα κερδίσουν περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ, Φοντάνα και μετά Ρούμπιχ. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνο και θα υποβάλω συγκεκριμένα ερωτήματα στον Επιτροπό που τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ. Εμεί ε, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο θέλαμε να υποβάλουμε ερωτήματα. Αναρωτιόμαστε για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη που έχουν περιφερειακή δομή, αν θα υπάρχουν κάποια συστήματα πριμοδότησης περιφερειών. Αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσε να γίνει στα κράτη εκείνη όπου υπάρχουν περιφέρειες που είναι ενάρετες σε σχέση με ένα κράτος που είναι λιγότερο ενάρετο από αυτή τη σκοπιά σε ό,τι αφορά την απόδοση και πώς θα μπορούσε να επιληθεί μια τέτοια σχετική κατάσταση. Αναρωτιόμασταν επίσης σε σχέση με, τις, ε, με το coupling ε, διαφόρων περιοχών, τι γίνεται με ευαίσθητα προϊόντα όπως είναι το γάλα ή ο καπνός. Ξέρουμε ότι η κατάσταση τέτοιου τύπου υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Και θα θέλαμε να μάθουμε επίσης σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ξέρουμε ότι τα προϊόντα μας, τα προϊόντα ποιότητας, που θέλουμε να φτάνουν στην αγορά πρέπει να εξετάζουμε πώς ακριβώς παράγονται και ποιο είναι το υπόδειγμα, το παραγωγικό μοντέλο και ποια θα είναι η πολιτική προώθηση τέτοιου είδους ποιοτικών προϊόντων. Και τέλος κύριε Επίτροπε, κάτι το οποίο κάθε φορά ε, σας θέτω όταν έρχεστε να μας ε, συζητήσετε Μιλήσατε για ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωση, και σίγουρα είναι κάτι θετικό να πραγματεύεστε το ζήτημα αυτό. Είναι όμω εξίσου αληθές ότι αν δεν ασχοληθούμε με αυτό που συμβαίνει και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση, αν ασχοληθούμε με τις εισαγωγέ που κάνουμε, Δυστυχώ, υπερβολικά συχνά προκαλώντα αθέμητο ανταγωνισμό έναντι των δικών μα προϊόντων, τότε απλώς πάντα θα κάνουμε το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή ποτέ θα καταφέρουμε να έχουμε ε, αηφόρο και βιώσιμη γεωργία για τους ε, ε, παραγωγούς μας. Εάν δεν δούμε και δεν υπάρχουν συμφωνίες, αν θέλετε, με το εισαγωγές από το Μαρόκο και δει πόσο πλήττουν τους Ισπανούς παραγωγούς, τι μπορούμε να κάνουμε σχέση με την παραγωγικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρούμπιξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την πολύ βαθιά μου ικανοποίηση για την συνάντηση αυτή. Πάντα χαίρομαι όταν έρχεστε και είναι πολύ καλό σημαντικό, πολύ ευχάριστο σημάδι ότι έρχεστε τόσο συχνά. Εκ μέρους της ομάδας μας προβληματιζόμαστε για πάρα πολλά θέματα αλλά ιδιαίτερα ε, μας ε, προβληματίζει το θέμα κοινωνικής ε, ανισότητας που διαφαίνεται από την αυτή πρόταση. Κάτι άλλο που επίσης προβληματίζει πάρα πολύ είναι η αύξηση του διοικητικού άχθους στους γεωργούς. Για να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν δικαίωμα και είναι δικαιούχοι σε οτιδήποτε θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλέ και πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα ήθελα να πω τώρα λίγα πράγματα για την Λετωνία. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος στους γεωργούς τη Βαλτική. Ε, και στην Εστονία και στη Λουθανία υπάρχει σχετικό πρόβλημα. Πάρα πολλοί ε, βουλευτές ε, του Ευρωκοινοβουλίου έχουν πάει να τους μιλήσουν και μας ζητούν να μετατρέψουμε τα λόγια μας σε πράξεις. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας. Θέλουμε κοινωνική προστασία, θέλουμε ισοτιμία, ισότιμο και νομότυπο ανταγωνισμό. Βλέποντας όμως την πράξη, βλέπουμε ότι οι βαλτικές χώρες και η Δήλη το 2020 θα λάβουν μόλις το 52% του μέσου κοινοτικού όρου σε άμεση πληρωμές. Αυτό δεν συνιστά ισότητα. Σίγουρα δεν είναι ίσες ευκαιρίες για την ανταγωνιστικότητα έτσι λοιπόν οι αγρότες μας θα πρέπει να πληθούν και να ζητήσουν τουλάχιστον ένα 90% άμεση προμές, τουλάχιστον στο 90% του μέσου κοινοτικού όρου το 2020. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές δαπάνες. Είναι ένα, μόλις ένα ποσό 2 δις για το σύνολο των βαλτικών χωρών για την επόμενη 7 αιτία που πρόκειται να τεθούν σε αμεση προ... γεωργικές προμές. Ελπίζω να ακουστεί εδώ η πρότασή μου και να επιτύχουμε αυτό που προσπαθούμε. Και σήμερα ο κ. Μπέζος, προ, πρόεδρος της Λετωνίας, είναι σε επίσημη επίσκεψη στις Βρυξέλλες και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα υποστηρίξει την πρόταση αυτή. Θα έχουμε κάποιο χρόνο να δουλέψουμε πάνω στην πρόταση αυτή, όμως η συγκεκριμένη αυτή έκθεση πραγματικά δεν είναι καθόλου προς ικανοποίηση των βαλτικών χωρών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα οι τρει ηγητέ. Όπω ξέρετε, ο Λουίς Κάπολαν Σαντό ε, Σάβολ Σαντέ και Λουζάνη Λαβία. Ο Λουί ε, παρατηρείται γιατί μίλησε προηγουμένω, οπότε δίνεται περισσότερη δυνατότητα στο Μισελ Νταντέν, Στεφάν Φολ. Ο Μισελ πρώτο. Ερχόμαστε σε αυτή την ε, δύσκολη αυτή άσκηση σε ό,τι που, που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε σχέση με αυτό που μας είπατε, συμφωνώ ότι η γεωργία θα πρέπει να συνδυάζει οικονομική αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντικές αποδόσεις σε ένα πλαίσιο πολύ, ε, πολύ έντονου και οξέως παγκόσμιου ανταγωνισμού. Το θέμα λοιπόν της ανταγωνιστικότητας είναι σημαντικό για να υπάρχει μια επαρκής ε, απόδοση στον τομέα και των τροφίμων και της γεωργίας. Θα πρέπει λοιπόν πραγματιστικοί και ρεαλιστικοί κανόνες για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της ανταγωνισμού. Η ενδυνάμωση των διαπαγγελματικών οργανώσεων και των ενώσεων των γεωργών που βρίσκεται αν θέλετε στα πλαίσια και στο περιθώριο του σχετικού δικαίου του ανταγωνιστικού θα δώσει τη δυνατότητα να είναι πιο ισχυρό ο γεωργό και να έχει ένα πολύ πιο ισότιμο μερίδιο τη προστιθέμενη αξία. Α μην ξεχνάμε ότι μιλάμε αφενός μεν για 13,5 ε, εκατομμύρια γεωργών και πέντε μεγάλους ε, ε, οίκους ε, ομίλους διανομής. Επομένως δεν πρέπει να εξαιρετηθούν οι γεωργικές οργανώσεις. Θα πρέπει οι γεωργικές οργανώσεις και οι επαγγελματικέ οργανώσεις να έχουν πραγματική εξουσία στα περιθώρια, αν θέλετε, τους, ε, τομέα αυτού που πρέπει να δουλέψουμε. Εάν θέλουμε διαχείριση των κρίσεων χωρίς να ξεκινούμε από τις βάσεις των διαφερομένων, έτσι όπως μας το παρουσιάσετε εσείς, θεωρώ τα προτινόμενα εργαλεία σε σχέση με τα εργαλεία τα οποία είχε προτείνει και τι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπολείπονται ακόμα σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητα απόδραση με μια σωστή διαχείριση των αγορών που φαίνεται λίγο να τι έχουμε ξεχάσει με την πρόταση αυτή. Γιατί αν κατάλαβα καλά, από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω διαβάζοντα και διαβάζω την πρόταση, πλέον επιβεβαιώνεται από την ε, η Επιτροπή ότι εγκαταλείπεται ε, η διαχείριση και ο διακανονισμός στον τομέα της κοινή οργάνωση των αγορών ε, αλλά και μια αναδιάρθρωση των τομέων ζάχαρης και ίνου θα πρέπει να έχουμε προσαρμογή στι προκλήσει του 21ου αιώνα. Αλλά η αναγκαιότητα αναγνωσιμότητα των οικονομικών επιταγών, ιδιαίτερα στο γεωρικό τομέα, μα υποχρεώνει να βρούμε όπου είναι δυνατόν ευέλικτα εργαλεία που θα μπορούν να εξασφαλίσουν και την απρόσκοπτη διατροφική, την ε, ευσυτιστική ε, παροχή, αλλά και την βιωσιμότητα γεωρικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την Ήπειρο. Υπό αυτή λοιπόν, τη σκοπιά θα ήθελα να δω την προτινόμενη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Ευχαριστούμε, Μισελ. Στάνλε Φόλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο όμως, χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ καταρχάς που ήρθατε εδώ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις απλές. Καταρχάς, η μάχη όσον αφορά τον προπολογισμό της ΚΑΠ δεν έχει κερδιθεί και χρειάζεται δέσμευση από όλους και συγκεκριμένα από εσά. Με ικανοποιεί αυτά που άκουσα από εσά ότι για κάποιες παραγωγές θα παραμένει το ελάχιστο κάπλινγκ και έχουμε κερδίσει στο Τρίτο, για το πρασίνισμα. Πιστεύω ότι οι προτάσεις τις οποίες κάνετε διατηρούν αυτό το οποίο υπάρχει, αλλά δεν ανοίγουν νέε προοπτικέ για νέα μοντέλα ανάπτυξης, τα οποία θα πρέπει να είναι ε, περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελεσματικά. Το να υπάρχει μία ε, αμυψισφορά, μία αγρανάπαυση, ένα μικρό βοσκοτόπου κτλ. Αυτά τα μέτρα δεν αρκούν για, για την καλύτερη χρήση των εδαφών τελευταίο πρόβλημα. Το είχα πει και όταν έγινε η ανακοίνωσή σας πριν από ένα χρόνο. Πιστεύω ότι όσον αφορά την ρύθμιση των αγορών, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή θα πρέπει να ε, διαχειριστούμε την προσφορά, χρειάζονται μέτρα. Χρειάζονται μέτρα τα οποία να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Βλέπετε πια πώς ε, διακυμαίνονται οι τιμές. Βλέπετε ότι υπάρχει κρίση στην κρίση. Τα μέτρα τα οποία έχουμε τώρα στη διάθεσή μας δεν μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Θα ήθελα να ξέρω ότι όσον αφορά το αποθεματικό της κρίσης που είχε προβλεφθεί υπάρχει εδώ στον κανονισμό. Μιλήσατε για 2-3 δις. Τι, ακριβώς, σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Επίσης, τελευταία παρατήρηση, θα πρέπει όσον αφορά την ε, ε, διατροφική ασφάλεια να την ρυθμίσουμε σε ένα επίπεδο ανώτερο από αυτό το οποίο αναφέρεται. Τζοβάν Λαβία και μετά ο, ο απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς ο οριζόντιος κανονισμός για τη διαχείριση και τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αφορά τα πάντα και όλο το σύστημα. Ήθελα να πω όμως ότι αυτό το οποίο είναι πιο σκοτεινό και πιο δύσκολο να καταλάβουμε στον γεωργικό τομέα, έστω και αν έχει μεγάλες συνέπειες, είναι ακριβώς ε, το κείμενο το οποίο μας παρουσιάστηκε σήμερα. Ε, ακούσαμε κάποια, κάποια στοιχεία βέβαια σήμερα, θα το διαβάσουμε με μεγαλύτερες ε, λεπτομέρειες και θα έχουμε το, την δυνατότητα μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ευθυγράμμισης με την, με την συνθήκη της Λισαβόνας να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε κάπως το κείμενο υπάρχει εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Κομισιόν που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας και προφανώς ε, ε, μεταρρυθμίζονται, αναδιαρθρώνονται οι σχέσεις ε, ανάμεσα στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Τώρα για τις δεσμεύσεις των πόρων εδώ έχει γίνει μια πρόταση που φαίνεται ότι προχωρούμε με ένα προοδευτικό σύστημα ενώ στην πρόταση η οποία, την οποία είχε υποβάλει η Κομισιόν μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ε, συνοχής τα πράγματα δεν ήταν ε, ακριβώς έτσι. Θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη τα οποία έχουν ε, πολύ ισχυρές περιφέρειες και κράτη τα οποία έχουν ένα κεντρικό, μια και πιο ισχυρή κεντρική δομή. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε. Η αναλογικότητα των ε, ελέγχων, ένα άλλο στοιχείο που είναι και αυτό σημαντικό, αλλά θα πρέπει να το ρυθμίσουμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Θα πρέπει, πιστεύω, να δούμε και κάποιες πτυχές που είναι σημαντικές, έστω και αν φαίνονται δευτερεύουσα σημασίες. Καταρχάς η εξακρίβωση από τους ε, κοινοτικούς οργάνους. Ποια είναι τα... Ε, ε, και, κοινοτικά όργανα, συγγνώμη. ποιο είναι το σχέδιο και το πλάνο ελέγχων και επιθεωρήσεων. Πώς θα δίνονται, πώς ποιος αναλαμβάνει τους ελέγχους αυτούς. Τώρα δεν θα πούμε σε λεπτομέρεια βέβαια, αλλά τέλος πάντων οι εξακριβώσεις ε, και η έλεγχη συμμόρφωσης. Ήδη ε, αποτέλεσε ένα αντικείμενο κριτικής από πλευρά του Ελεκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για, τους, για τις καταποκοπήν μειώσεις κτλ. Ήδη ασκήθηκε κριτική από την Κομισιόν διότι υιοθετήθηκαν στο 90% των περιπτώσεων. Θα πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά και να δούμε στη νέα πρόταση πόσες από αυτές τι τις που ασκήθηκαν από το Ελεκτικό Συνέδριο έχουν ληφθεί υπόψη από την Κομισιό. Ευχαριστώ Τζοβάνι. Νομίζω κύριε Επίτροπε εμείς σεβαστήκαμε το χρόνο. Έχετε την δυνατότητα ε, να απαντήσετε ε, και να πω και στους συναδέλφους, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος εδώ ομιλητών, ότι με το γραφείο του, του Επιτρόπου ε, έτσι ώστε να δώσουμε όλες τις παρεμβάσεις στο γραφείο και να μας ε, δοθεί απάντηση. Ευχαριστώ πάλι. Προσπαθήσω να παραμείνω ακριβώς στη ζήτηση αυτή, το γνωρίζεις, μέχρι τη στιγμή που θα συνήθως μένω μέχρι ότου ο καθένας μπορεί να ε, λάβει το λόγο. Τώρα πρέπει να κάνουμε συμβασμό μεταξύ της ταχύτητας παρουσίας εδώ, που αφορά και σας και εμένα, και του, περιορισμού, του χρονικού περιορισμού που υπάρχει. Αλλά όπως είπε ο Παύλο, σας δίνω την υπόσχεση να επανέλθω όσες φορές κρυθεί απαραίτητο για να υπάρξει μια ει και κατ' συζήτηση για όλες τις προτάσεις. Ε, εντάχει λοιπόν κάποιε πρώτε αντιδράσεις στις ε, πρώτα ερωτήματα και παρατηρήσει σα. Ε, συνολικά σε ό,τι αφορά το γραφειοκρατικό άχθος. Νομίζω ότι το είπαμε κατά επανάληψη. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα πλαίσια μιας ΚΑΠ. Μιλάω για την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της. Μεταξύ σε μια διελκυστίδα αφενός μεν των αναγκών του να υπάρξουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα, αλλά και να υπάρξει απλούστευση. Και πρέπει να βρούμε τον, ε, τη μέση οδό, ώστε να έχουμε την απλούστε δυνατή διαδικασία, αλλά και να έχουμε και τα περισσότερα και καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γιατί η δημόσια πολιτική μετράται επίση και με την ικανότητα κατάδειξη ε, αποτελεσμάτων. Το απλούστερο θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα, δηλαδή να δίνουμε τα χρήματα χωρί να ζητάμε τίποτα σε αντιστάθμισμα. Θα ήταν το απλούστερο. Νομίζω και θα συμφωνείτε μαζί μου δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να ζητάμε πράγματα που θα δίνουν αποτελέσματα, χωρίς όμως να είναι πολύπλοκος ο τρόπο. Αυτή είναι η κατευθυντήρια γραμμή που μας οδηγεί όταν συζητήσαμε και για τα μέτρα ε, πρασινίσματος. Να είναι μέτρα απλά και ελέγξιμα. Το είχαμε αυτό και στην ανακοίνηση. Το υπενθυμίζω, σας υπενθυμίζω ότι το πράσινη κάλυψη εδαφών που είχαμε προτείνει, μετά από μια σχετική μελέτη επιπτώσεων, είδαμε ότι αυτό το μέτρο μπορεί να προκαλούσε επιπρόσθετες ε, γραφειοκρατικές ε, διαδικασίες και ελέγχους και γι' αυτό και την απορρίψαμε εκείνη την πρόταση και προτείναμε κάτι άλλο απλούστερο ίσως προτείναμε κάποια μέτρα όχι τόσο φιλόδοξα για κάποιους ή υπερβολικά φιλόδοξα για άλλους, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθήσαμε να βρούμε τον απλούστερο δυνατό τρόπο χωρίς βέβαια αυτό, αυτό να συνεπάγεται επιπρόσθετο κόστος για τους γεωργούς. Μιλούσατε για το 7% της αγρανόπαυσης. Δεν είναι 7% η αγρανόπαυση, γιατί το 7% των εδαφών αυτών μπορεί να παίρνει κάποιες μορφές ε, ε, βλάστησης που κρατά τα εδάφη γόνιμα, ακόμα και αν δεν καλλιεργούνται για παραγωγικούς λόγους και που αυτή τη στιγμή δεν είναι ε, επιλέξιμα για πληρωμές. Μπορεί να μην είναι επιλέξιμα για γεωργικές πληρωμές, αλλά τα κρατάει ο αγρότης σε βλάστηση. Έχουμε τις λεγόμενες ε, ε, δασικές, ε, δασικά πετάσματα, δασικές ε, ζώνες δηλαδή. Έχουμε αυτές τις ζώνες ε, με δέντρα που θα είναι επίσης επιλέξιμα μέσα σε αυτό το 7%. Υπάρχουν επίσης μορφές βλάστησης που είναι χρήσιμες για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων. Ακόμα και δεν είναι άμεσα παραγωγικές που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το 7% για τις ε, ε, διπλές, για τις ε, πληρωμές coupling διατηρηθήκαν, αλλά με την ε, διευκρίνηση ότι θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο ώστε να είναι αιτιολογημένη η χρήση αυτή, ώστε να κρατήσουμε τον προσανατολισμό προς την αγορά, αλλά συγκεκριμένε περιστάσεις. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο το αιτιολογεί. Σε ό,τι αφορά την σύγκληση, γνωρίζω πολύ καλά το πρόβλημα των βαλτικών χωρών και το γεγονός ότι η παρούσα πρόταση δεν είναι ίσως τόσο φιλόδοξη σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν ε, οι συμπολίτες της Βαλτικής και ίσως με τους στόχους που είχα εγώ από την αρχή. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια της Realpolitik, όντας πραγματιστές. Είναι πρώτη φορά που η ΚΑΠ και ο προπολογισμό της ε, αποφασίζονται εν παραλίλω με, με όλη μεταρρύθμιση που επέρχεται. Έχει και άλλες συνιστώσεις ε, του προπολογισμού η κοινή αγροτική πολιτική και πιστεύω ότι θα υπάρξουν θέματα προς συζήτηση και ίσως δοθούν συγκεκριμένες λύσεις που θα, ξεπεράσουν το σχετικό και το πολύ απλό ε, πλαίσιο της κοινή αγροτικής πολιτικής. Σας υπενθυμίζω αυτόν τον περιορισμό του 30% της διαφοράς, το 1 τρίτον δηλαδή της διαφοράς είχε ήδη αποφασιστεί στην Επιτροπή μέσα στις δημοσιονομικές προοπτικές, όχι στην ΚΑΠ. Βλέπετε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που ξεπερνά την απλή κοινή αγροτική πολιτική, γιατί πρόκειται και για ένα δημοσιονομικό μοίρασμα μεταξύ των κρατών μελών που εντάσσονται και σε άλλε γραμμέ του προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τον ε, κανονισμό τη παραγωγή, είπαμε και προηγουμένω ότι τα μέτρα τη αγορά θα πρέπει να εξασφαλίζουν πραγματική επιστηστική ασφάλεια. Αυτό προτείναμε. Υπάρχουν μέτρα, τομεακά μέτρα οργάνωση τη αγορά, πριν από λίγα χρόνια πέρασαν με κάποιε συγκεκριμένε όπω για τον τομέα του ίνου και των απορροκυπευτικών. Κάναμε κάποιες προτάσεις για τον τομέα των γαλακτοκομικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει με εκθέσεις και προτάσεις το 2012-2013 και για τον ίνο και για τα απορροκυπευτικά. Είναι, είναι μηχανισμοί συγκεκριμένοι που θέλουμε να διατηρήσουμε, αλλά αυτό το οποίο προτείνει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το νομοθετικό πακέτο είναι ε, νομοθετικές προτάσεις γενικής τάξης για να υπάρχει ακριβώς δίκτυα ασφαλείας που θα μπορεί να κινητοποιείται άμεσα και με ασφάλεια. Νομίζω ότι έχετε σχετικές ε, προτάσεις να υποβάλλετε μεταξύ ε, που μπορείτε να μελετήσετε και που έχουν υποβληθεί. Ε, εξάλλου, σε ό,τι αφορά την οργάνωση των αγορών θα πρέπει να είναι σαφές κλειδί για κάθε διαχείριση κρίσης, κάθε φύσης. Νομίζω ότι για να είμαστε απλούστερα δυνατόν, χωρί γραφειοκρατία και να λειτουργούμε το συντομότερο δυνατόν και στην πηγή του θέματο, είναι η οργάνωση των παραγωγών που πρέπει να ενισχυθούν και να του δώσουμε πραγματικά τα μέσα για να μπορέσουν να δράσουν. Προ αυτή την κατεύθυνση λοιπόν σα προτείνουμε να δουλέψουμε και αν μπορούμε να ενισχύσουμε κάποια στοιχεία θα τα συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ε, είμαι πεπισμένο ότι με αυτή τη διαδικασία λήψη αποφάσεων δεν βρισκόμαστε κατά στο 2003, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 15 κράτη-μέλη κλείνοντα σε μια αίθουσα για μια μισή μέρα για να πάρουν τι τελικέ αποφάσει. Θα είναι πολύ μακροπρόθεση, πιο, μακρο, μακρόπνοη αυτή η προσπάθεια συνεργασία, ανάλυση των κειμένων, ε, σύνθεση και συγκυρισμού προτάσεων, προτάσεων που έχετε ήδη υπό εξέταση, και ο, και ίδιος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το πραγματικό παιχνίδι της ε, ενεργού συμμετοχικής δημοκρατίας και υπό αυτό το πνεύμα παρουσιάζω το κείμενο αυτό και υπό αυτό το πνεύμα θα επανέλθω ε, σύντομα τις επόμενες μέρες και επόμενες εβδομάδες. Και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με προσκαλέσατε και με δεχθήκατε σήμερα.